Αρχίζουμε. Σημείο 9 στην ημερήσια διάταξη. Καλωσορίζουμε εδώ την Υπουργό Νάτια Καλβίνιο, Υπουργό Οικονομίας και Απασχόλησης της Ισπανίας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε για αυτό τον οικονομικό διάλογο μαζί σας με την Ισπανία. Και ξέρετε ότι κυρία Καλβίνιο έχει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο γιατί είναι υπεύθυνη και για την ε, κυβερνητική επιτροπή όπου εκεί μαζεύονται όλοι οι υπουργοί. Οπότε ξέρει και από Eurogroup και Ecofin και θα μας μιλήσει και για διάφορα ζητήματα που απασχολούν τη δικιά μας επιτροπή. Ό,τι ανακοινώσει έχω θα σας τις κάνω μετά. Είμαστε λοιπόν στον οικονομικό διάλογο αυτόν με την Ισπανία. Όπως γνωρίζετε, η Ισπανία έχει θετικές προοπτικές. Και παρουσίασε έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό Επικεντρωμένο πολύ στις κοινωνικές δαπάνες, τη συνοχή, την καινοτομία και τις επενδύσεις. Θα μας μιλήσει για όλα αυτά σίγουρα η κυρία Καλβίνιο. Επίσης, αλλά και θα συζητήσουμε μετά, ε, θα μας πει και για τα ισπανικά ζητήματα, αλλά και γενικότερα ευρωπαϊκά. Για την ευάθυση στην ΟΝΕ, μια διαδικασία που όπως γνωρίζετε είναι ζωτική σημασία και για μας. Δουλεύουμε και εμείς πάνω στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλουμε να ξέρουμε τις απόψεις σας και για αυτό το θέμα και για τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης, να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Σίγουρα οι συγητές μας ενδιαφέρονται πολύ. Εσείς λοιπόν τώρα έχετε το λόγο. Θα ακούσουμε τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις και στη συνέχεια, όπως κάνουμε συνήθως, θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις. Υπουργό, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Γουαλτιέρη. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ τη Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που μου δίνεται ευκαιρία αυτή να έρθω εδώ στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για χρόνια η Επιτροπή αυτή έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μου ζωή εξακολουθώ να έχω πολλούς φίλους από την Επιτροπή σας. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που για πρώτη φορά βρίσκομαι εδώ ω υπουργό ε, Οικονομίας τη Ισπανία. Οπότε πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή που μου δώσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Επιπλέον, η συνάντηση αυτή εδώ λαμβάνει χώρα σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή όπως το ακούσαμε. Όταν η, Ισπανική κυβέρνηση παρουσίασε το νομοσχέδιο για τον προπολογισμό της χώρας για το 2019, όπου αντικατοπτρίζονται οι οικονομικές μας προτεραιότητες. Πρόκειται για ένα σχέδιο προπολογισμού που προβλέπει η οικονομική ανάπτυξη στην Ισπανία, ότι θα διατηρηθεί και το 2019, με δείκτες που ε, ξεπερνούν από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Θα είναι παραπάνω λοιπόν από ότι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πολλές άλλες αναπτυγμένες χώρες. Πρόκειται για ένα σχέδιο προπολογισμού που περιλαμβάνει τους τρεις πυλώνες της δικιάς μας οικονομικής πολιτικής, στους οποίους και θα αναφερθώ στη συνέχεια, αλλά που συνοψίζονται ως εξής. Πρώτον, δεσμευόμαστε για δημοσιονομική πειθαρχία. Ο στόχος μας για το δημόσιο έλλειμμα για το 2019 είναι 1,3% του ΕΠ. Ενώ 2,7% φαίνεται ότι κλείνει το 2018. Για πρώτη φορά το 2019 πετυχαίνουμε επίσης πρωτογενές πλεόνασμα. Και έτσι μπορούμε να αρχίζουμε να διορθώνουμε μία από τις πιο σημαντικές ανισορροπίες που κληρονομήσαμε από την κρίση, που είναι το μεγάλο δημόσιο χρέος και η αναλογία του δημοσίου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας. Δεύτερος πυλώνας της οικονομικής μας πολιτικής είναι ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στην κοινωνική συνοχή Αναφέρθηκε σε αυτό πριν από λίγο κύριος ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη. Και υιοθετούμε ειδικά μέτρα ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να υποφεληθούν από την ανάπτυξη. Να θέλουμε να μειώσουμε τις ανισότητες και να συνεισφέρουμε στην κοινωνική βιωσιμότητα. Κάτι το οποίο είναι αναγκαίο αν θέλουμε να έχουμε οικονομική ε, επίση βιωσιμότητα. Και ο τρίτος πυλώνας είναι ότι Θέλουμε να προχωρήσουμε τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα της χώρας μας και να ετοιμαστούμε για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ετοιμάζουμε επίσης το λεγόμενη Agenda for Change. Είναι η στόχη μας για την αλλαγή όπου συμπεριλαμβάνονται οι στόχοι μας που θεωρούμε ότι είναι αναγκαίοι για να πετύχουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Και πριν συνεχίσω, για την οικονομική μας πολιτική, επιτρέψτε μου να σας δώσω λιγάκι το οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Ξεκινάω από την παγκόσμια οικονομία. Όλες οι προβλέψεις λένε ότι η οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίω θα συνεχίσει θετικά αυτή τη χρονιά. Λιγότερο όμως με λιγότερη ένταση και θα υπάρχουν και διαφορές ανάμεσα στις περιφέρειες και τις χώρες του κόσμου. Πολύ περισσότερο από ό,τι παλιότερα ελοχεύουν κίνδυνοι και αβεβαιότητα με επιπτώσεις που θα φανούν κατά τη διάρκεια του 2019. Δεν χρειάζεται εγώ να σας εξηγήσω όλα αυτά, τα γνωρίζετε φυσικά, τα συζητάτε κάθε μέρα. Και έτσι θα διαμορφωθούν και οι διάφορες προκλήσεις που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην Ευρωζώνη το 2019 οι προβλέψεις έχουν ε, πέσει κάπως. Και νομίζω ότι πρέπει να πιεστούμε όλοι περισσότερο ώστε να προχωρήσουμε στην ευάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθω σε λίγο. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν η ισπανική οικονομία έχει ένα σημαντικό δίκτυ ανάπτυξης που θα διατηρηθεί και το 2019 ελπίζουμε. Η πρόβλεψή μας είναι της τάξης του 2,6% το 2018 και 2,2% το 2019. Πρόκειται για δείκτες σημαντικούς οι οποίοι βέβαια έχουν πέσει σε σχέση με το 2015 εξαιτία ε, του κύκλου στον οποίο βρισκόμαστε. Αλλά παραμένουν πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Επίσης, όσον αφορά το ΕΠΑ, το μοντέλο ανάπτυξη στην Ισπανία είναι πιο ισορροπημένο από τις άλλους κύκλους της ιστορίας μας. Έχει υπάρξει μεγάλη αύξηση στην απασχόληση. 3% ε, το 2018, που σημαίνει ότι μειώθηκε η ανεργία κατά 6% περίπου πέρυσι. Επιπλέον αυτή η οικονομική ανάπτυξη συνοδεύεται και από πλεόνασμα στους τρέχοντες λογαριασμούς που είναι κάτι καινούριο και σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. παρά το μεγάλο ε, εξωτερικό χρέος που έχουμε και που κληρονομήσαμε επίσης από την κρίση. Συνεχίζουμε λοιπόν να βγαίνουμε από την τελμάτωση. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο οικονομικό που θα πρέπει να είναι ευνοϊκό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να προχωρήσουμε βάσει των τριών πυλώνων που σας παρουσίασα πριν. Πρώτα απ' όλα, δημοσιονομική πειθαρχία. Σας είπα ότι είναι ένα στοιχείο πολύ βασικό για το σχέδια της κυβέρνησης. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με τη μείωση του ελλείμματος, να μειώσουμε και το χρέος και Συνεχίζοντας έτσι, μπορούμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των οικονομικών ε, αγορών που ήδη έχουν δείξει απέναντι στην ισπανική οικονομία. Ήδη το 2018, παρά τις διάφορες αβεβαιότητες, η κατάσταση ήταν ε, θετική όσον αφορά τις επενδύσεις στο δημόσιο τομέα. Και στις αρχές του 2019 φαίνεται ότι τα πράγματα είναι επίσης πολύ ε, ευνοϊκά. Οι διάφορες δημόσιες προσφορές που έχουν γίνει, έχω εδώ μαζί μου και τον Γενικό Γραμματέα ο οποίος ε, μπορεί να το επιβεβαιώσει πόσο θετική είναι η κατάσταση. Οι δημόσιες προσφορές λοιπόν που έχουμε κάνει μέχρι τώρα έχουν πολύ καλά αποτελέσματα ρεκόρ και μας επιτρέπουν να μειώσουμε ε, το κόστος της χρηματοδότησης του ισπανικού χρέους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την κυβέρνησή μας γιατί κάθε χρόνο πρέπει κάπου 30 δισευρώ να δίνουμε για την εξυπηρέτηση αυτή κάτι το οποίο θα ήταν πολύ πιο παραγωγικό αν μπορούσε να πάει στην εκπαίδευση, στην υγεία ή στην καινοτομία και την ανάπτυξη. Η εμπιστοσύνη λοιπόν των οικονομικών αγορών είναι κάτι αναγκαίο. Αυτό το μάθαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης και αυτό ακριβώ και εξηγεί και τον πρώτο πυλώνα βιωσιμότητας του προγράμματος της κυβέρνησης. Όμω επίση χρειαζόμαστε και την εμπιστοσύνη των πολιτών και γι' αυτό έρχομαι στο δεύτερο πυλώνα που είναι το στίχημα που έχουμε βάλει υπέρ τη κοινωνικής συνοχής. Γιατί η δημοσιονομική πειθαρχία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σαν άλοθη για να μην λύνουμε το βασικό πρόβλημα της χώρας που είναι η μεγάλη αύξηση των ανισοτήτων που είχαμε μετά από την οικονομική κρίση. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε η οικονομική ανάπτυξη να αγγίξει και τον τελευταίο πολίτη. Θέλουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης με συμμετοχή όλων, χωρίς αποκλεισμούς. Και αυτό τονίζουν και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι διάφοροι διεθνεί οργανισμοί και είμαστε και εμεί πεπισμένοι γι' αυτό και στο σχέδιο προπολογισμού που στείλαμε και εμεί ε, στο Ισπανικό Κοινοβούλιο συμπεριλαμβάνεται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, το πιο φιλόδοξο δυνατό στα πλαίσια τη δημοσιονομική πειθαρχία υπέρ κοινωνικών πολιτικών. Εκπαίδευση για τα παιδιά 0 έω 3 ετών αύξηση του ελάχιστου μισθού, ε, των συντάξεων, κοινωνική πολιτική υπέρ της οικογένειας, για να βοηθήσουμε κυρίως τους πιο ευάλωτους πολίτες. Πρόκειται για στόχους και για ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας επιτρέψει να λύσουμε το πρόβλημα των ε, ανισορροπιών, των ανισοτήτων που έχουμε. Ο τρίτος πυλώνας των οικονομικών μας στόχο είναι για να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικέ προκλήσεις. Βασιζόμαστε σε μια βιώσιμη ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα, βιώσιμη οικονομικά, βιώσιμη κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα άρχισε να δουλεύει για να υπάρξει συντονισμός ανάμεσα στα διάφορα υπουργεία. Το ανέφερε αυτό ο κ. Γκουαλτιέρη πριν για να προχωρήσουμε ε, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, εκπαίδευση, με το ανθρώπινο δυναμικό και την ε, κατάρτιση, να στηρίξουμε την μετάβαση, την οικολογική μετάβαση, όπως επίσης και την τεχνολογική και ψηφιακή να εγγυθούμε τις ε, ψηφιακές ε, τεχνολογίες, να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες και να έχουμε και μια δικητική δομή, μια δίκηση η οποία να είναι πιο αποτελεσματική και να εξυπηρετεί τον πολίτη. Προκειμένου αυτή η σταθερότητα να διατηρηθεί και στο μέλλον, είναι αναγκαίο η Ευρωζώνη, το ενιαίο μας νόμισμα, το ευρώ, να αποτελεί πηγή σταθερότητας και εμπιστοσύνης. Και γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ βασικό να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας πραγματικής οικονομικής και νομισματικής ένωσης, γιατί τότε θα είμαστε όλοι πιο δυνατοί και καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Όπως όλοι γνωρίζετε, το Eurogroup το προηγούμενο μήνα κατέληξε σε συμφωνία για ένα πακέτο μέτρων που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία ενός δικτύου δημοσιονομικής ασφάλειας ενίσχυση επίσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του ESM, ε, αποφάσισε για προγράμματα εγγυήσεων στην περίπτωση που υπάρχει οικονομική αστάθεια και δημόσιο χρέος. Όλα αυτά είναι θετικές εξελίξεις που πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και πιστεύουμε ότι θα προχωρήσουμε γρήγορα αυτό το εξάμεινο. Σήμερα το πρωί, μάλλον χτες και σήμερα το πρωί στο Eurogroup και σήμερα και στο ECOFIN, βλέπουμε ότι υπάρχει μια στέρεα βάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Του επόμενου μήνε όμως πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Θέλουμε προδευτικά να δημιουργηθεί ε, αυτό το σύστημα αγγίσεων καταθέσεων, το ΕΝΤΙΣ. Η πρόταση αυτή βρίσκεται στο τραπέζι εδώ και πολύ καιρό. Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες που συνέχισε να ζητάει όθηση για να προχωρήσουμε και να ολοκληρωθεί αυτό το σύστημα, να έχουμε μία βάση ώστε να γίνουν στη συνέχεια οι πολιτικές συζητήσεις. Και επιπλέον, κάτι άλλο βασικό είναι η δημιουργία ενός προπολογισμού για την Ευρωζώνη, που να συμπεριλαμβάνει και μια λειτουργία σταθεροποίησης της Ευρωζώνης, για να έχουμε μια κοινή δημοσιονομική ικανότητα που να μπορεί να βοηθήσει σε περίπτωση ασυμμετρικών ε, σοκ και να μπορέσει να μας προστατεύσει από μια μελλοντική κρίση. Η... Το κοινό νόμισμα σημαίνει ότι παρετούμαστε από κάποια πράγματα εμείς που αποφασίζουμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το εργαλείο σταθεροποίησης ε, πιστεύουμε ότι πρέπει να λάβει υπόψη του πρώτα απ' όλα τους πολίτες, τους ανθρώπους. Και γι' αυτό εμείς επιμένουμε να υπάρχει ένας μηχανισμός που να έχει να κάνει με την εγγύηση στην απασχόληση. Μιλάμε τα τελευταία χρόνια για backstop, για τις αγορές, για τους επενδυτές. Να υπάρχει και ένα backstop, ένα δίκτυο ασφάλειας και για τους πολίτες, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Γιατί το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν είναι μόνο ε, για τα οικονομικά ζητήματα, είναι για τους ανθρώπους πρώτα απ' όλα. Οπότε για μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η μεταρρυθμιστική προσέγγιση. Και όπως είπε ο Πέντρο Σάντσες, ο πρόεδρος της κυβέρνησης της Ισπανίας πριν από λίγες μέρες στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, οι επόμενες ευρωεκλογέ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτούς που δεν πιστεύουν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και είναι δικιά μας ευθύνη να προστατεύσουμε την Ευρώπη προκειμένου η Ευρώπη να μπορέσει να συνεχίσει να κάνει αυτό που έκανε τις τελευταίες δεκαετίες ολοκλήρωσης, δηλαδή να προστατεύει εμάς τους πολίτες. Πρέπει να προχωρήσουμε για μια Ευρώπη πιο κοινωνική αλλά και να εμβαθύνουμε περισσότερο στην οικονομική και νομισματική πολιτική για να ελαχιστοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τις πιθανότητες να οδηγηθούμε σε μια νέα κρίση ή να μπορέσουμε να διορθώσουμε ό,τι επιπτώσεις μπορεί να έχει μια τέτοια μελλοντική κρίση. Αυτή είναι η στόχη μα λοιπόν σε εθνικό επίπεδο αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι φιλόδοξη σίγουρα όλη αυτή η στόχη. Η Ισπανία όμω είναι μια ισχυρή χώρα με μια κοινωνία που αντιστέκεται και με μια ιστορία γεμάτη επιτυχίε κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μια πρόκληση. Μετά από την τελευταία κρίση καταφέραμε να έχουμε πέντε χρόνια συνεχή ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων απασχόληση, πλεόνασμα στου τρέχοντε λογαριασμού και όλα αυτά τα πετύχαμε μειώνοντας τις ανισορροπίες. Και από πλευρά τη κυβέρνηση και τη ισπανική κοινωνία είμαστε αποφασισμένοι να υποφεληθούμε από την θετική οικονομική συγκυρία, ώστε η χώρα μα να βρεθεί στην καλύτερη δυνατό θέση για το μέλλον, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε υγιή δημοσιονομικά με την δημοσιονομική πειθαρχία δεσμευόμενοι όμως υπέρ μιας κοινωνικής ατζέντα για τους πολίτες μας, τους πιο ευάλωτους κυρίως, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να συμμετέχουν στην ανάπτυξη. Και έχουμε και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται η ισπανική οικονομία τα επόμενα χρόνια. Στη διαδικασία αυτή, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, όπως πάντα, θα δράσουμε ως ένα πιστός εταίρος ε, φιλόδοξος και επικοδομητικός υπέρ του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, Αγαπητοί Υπουργέ, για την πολύ σημαντική σας δήλωση και για την σαφή εικόνα που μας δώσετε για τον ισπανικό προπολογισμό και τις πολιτικές που στόχο έχουν την ευάθυνση της ε, νομισματικής ένωσης. Ε, πολύ μου άρεσε αυτό που είπατε ότι είναι όλα αυτά για τον κόσμο και τώρα πρώτα ο κύριος Γκαμπριέλ Μάτο από το ΕΛΚ. Ε, μπορώ και εγώ να χρησιμοποιήσω το χρόνο του ΕΛΚ, οπότε θα είμαστε ε, ε, εντάξει με τους χρόνους σας. Ευχαριστώ που ήρθατε. Στις προηγούμενες σας ε, καθήκοντα είχατε πολύ διαφορετική αποστολή από αυτή που έχετε σήμερα ως υπουργό της κυβέρνησης της Ισπανίας. Μπορώ να μοιραστώ πολλά μαζί σας, ε, να συμφωνήσω με πολλά από αυτά που είπατε, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, ανάπτυξη ή το χρέος. Ε, όμως άλλο είναι η θεωρία και άλλο είναι η πρακτική. Η πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου, και η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ε, δεν είναι ε, σωστή ε, κατά τη γνώμη μου. Προχωρά προς την αντίθετη μάλιστα κατεύθυνση. Είπατε πέντε χρόνια ανάπτυξης. Αν δεν ήταν το ΕΛΚ πριν θα σας έλεγα ότι ήταν χάρη στην προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό θα είχατε πει. Τώρα στους επόμενους έξι μήνες θα δούμε τι θα κάνει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Μιλήσατε όμως για στόχο μείωσης του χρέους ε, στο 95,4%. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκεκριμένη μέτρηση 96,2. Εσείς επίσης μιλάτε για κάποιους λογαριασμούς οι οποίοι πως είναι αμφισβητήσιμοι. Και δεν το λέω εγώ. Το λέει και η εφημερίδα El País που είναι αξιόπιστη εφημερίδα. Λέει λοιπόν πως ε, το δημόσιο χρέος θα είναι περίπου 2% και όχι 1,3% όπως ε, είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η Τράπεζα της Ισπανίας το Δεκέμβριο μείωναν τις προβλέψεις για ανάπτυξη ε, σε σχέση με τις αρχικές. Δεν είναι ιδανική δηλαδή η κατάσταση. Επίσης μας μιλήσατε για απασχόληση και είναι αλήθεια ότι δημιουργήθηκε πολλή απασχόληση στην Ισπανία. Δυστυχώς όμως ε, ε, επιβραδύνεται αυτή η κατάσταση και ε, δυστυχώς το 2018 δημιουργήθηκαν λιγότερες θέσεις απασχόλησης και προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν και λιγότερες το 19. Χρειάζονται λοιπόν μεταρρυθμίσει που δεν είναι εύκολο να γίνουν, αυτό αναμφίβολα, κυρίω με μια κυβέρνηση που δεν έχει πολύ ε, κοινοβουλευτική στήριξη και γι' αυτό θα θέλαμε να γνωρίζουμε Ακούσαμε για την εργατική μεταρρύθμιση. Ε, όμως εσείς ίδια είπατε πως αυτό το σύστημα μέχρι στιγμής λειτουργούσε πολύ καλά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Να κάνω, να κάνω και τους δύο γύρους παρέμβαση σε μία φορά. Αν δεν σας πειράζει, Πρόεδρε. Ναι, εντάξει, εντάξει. Καινοτομήσατε, αλλά δέχομαι την καινοτομία σας. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Και όσον αφορά τις εισαγωγέ. και τις, εξαγω... εξαγωγές μάλλον αυτές μειώθηκαν ε, ενώ είχαμε ε, αύξηση 1,3, τέσσερις φορές λιγότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο. και μπορούμε να πούμε διάφορα πράγματα για τη θέση που θα μπορούσαμε να έχουμε στην Ευρώπη. Τώρα όσο για τον προπολογισμό, όσον αφορά την κοινωνική συνοχή, νομίζω πως είναι πολύ θετικά αυτά που είπατε ότι δηλαδή η λιτότητα δεν πρέπει να είναι η δικαιολογία για να περικόπτονται οι κοινωνικές πολιτικές. Βεβαίως, αυτό που είναι όμως επίσης ε, σίγουρο είναι ότι τα έσοδα και οι δαπάνες θα πρέπει να, να ισοσκελίζονται και άρα θα πρέπει να βρεθούν κάποια έσοδα που να συμφωνούν με αυτά που προτίθεστε να δαπανίσετε. Όπως μου είπαν οι μου, υπάρχει διαφορά 29 περίπου ε, εκατομμυρίων. Πού θα, πώς θα καλυφθούν αυτά. Νομίζετε πως η Κομισιόν μπορεί πραγματικά να δεχτεί αυτό τον προϋπολογισμό που δεν είναι απόλυτα ισοσκελισμένος. Εντάξει, τώρα ξεπεράσατε όμως και το δεύτερο σας παρέμβαση, το χρόνο της δεύτερης σας παρέμβαση, διακόπτει ο Πρόεδρος. Εντάξει, εντάξει, σταματώ εδώ, στην ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μάτο. Ένα σωρό ερωτήσεις ε, μου θέσατε βέβαια. Και εγώ θα πρέπει να καταναλώσω διπλάσιο χρόνο για να μπορέσω να σας απαντήσω. Καταρχάς σας ευχαριστώ γιατί συμφωνήσατε με τους βασικούς στόχους όσον αφορά την ε, δημοσιονομική εξυγίανση. Ε, και αυτό δεν με εντυπωσιάζει γιατί σας υποβάλαμε έναν ε, προϋπολογισμό όπως τον είχε προτείνει και το δικό σας κόμμα με στόχο για έλλειμμα το 1,3% και αυτό προσπαθούμε να τηρήσουμε. Αυτό είναι ο στόχος ε, με τον οποίο υποβάλαμε αυτό το πρόγραμμα και για το οποίο έχουμε δεσμευθεί. Ελπίζω λοιπόν πως το ΠΠΕ θα στηρίξει αυτούς τους στόχους και αυτούς τους στόχους δηλαδή που η δική σας κυβέρνηση είχε θέσει επιτάπητος. Το ίδιο συμβαίνει και με τα προγράμματα για τις νέους φόρους. Ας πούμε, το ψηφιακό φόρος είχε ήδη προταθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, ακολουθεί το κοινοτικό μοντέλο, ακολουθεί τις χώρες που ε, πίεσαν για την επιβολή ε, κοινοτικού ψηφιακού φόρου και άρα πρόκειται για ένα νομοσχέδιο ε, που ελπίζω πως ε, θα βρει και τη στήριξη του ΠΕΠΕ στο ε, Ισπανική Βουλή. Τώρα κάποιοι γενικοί προβληματισμοί. Πρώτον, Ποια είναι η δυναμική και η εξέλιξη της χώρας μας σε αυτό το θέμα της ε, δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ε, θα πρέπει να σας πω ότι οι διάφορες κυβερνήσεις έχουν ε, προσπαθήσει, αλλά η πρόοδος ήταν αργή τα τελευταία χρόνια. Υπήρχαν κάποια χρόνια μεγαλύτερης οικονομικής ανάπτυξης, αλλά δεν το εκμεταλλευτήκαμε για να κάνουμε μια πραγματική ε, προσαρμογή το χρέος ήταν 100% του ΑΕΠ και δεν έχει μειωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Εμείς έχουμε έναν φιλόδοξο στόχο να μειώσουμε με διπλάσιο ρυθμό την αναλογία ε, του δημοσίου χρέου σε σχέση με το ΑΕΠ μέσα στον ε, επόμενο χρόνο θεωρούμε, όπως είπα και νωρίτερα, πως αυτός θα πρέπει να είναι ο κύριος στόχος από την άποψη της δημοσιονομικής πολιτικής. Και είναι αλήθεια πως οι αγορές δείχνουν εμπιστοσύνη και στήριξη σε αυτή τη στρατηγική, όπως σας έλεγα, όχι μόνο στη διάρκεια της ναι, εξαμήνου σοσιαλιστικής διακυβέρνησης τη χρήση του 18, αλλά και στις πρώτες εβδομάδες του τρέχοντος έτους, όπου βλέπουμε μέγα ενδιαφέρον και μεγάλη στήριξη σε αυτό το σενάριο μείωσης του δημόσιου χρέους. Υπάρχουν και κάποιες προβλέξεις ε, ε, για το έλλειμμα από πλευράς δημοσίων ε, και διεθνών οργανισμών. Αυτό δεν εντυπωσιάζει βέβαια, όπως όλοι γνωρίζετε πολύ καλά. Ε, ακόμα και όταν είναι τέσσερις μόνο οικονομολόγοι συγκεντρωμένοι, επικρατούν πέντε διαφορετικές απόψεις. Άρα για την κυβέρνησή μας αυτό το οποίο επιλέξαμε είναι να είμαστε συνετοί και πολύ προσεκτικοί. Ε, έχουμε λοιπόν ακολουθήσει τις πιο ε, συγκρατημένες προβλέψεις όσον αφορά την ανάπτυξη, την αύξηση των τιμών, την τιμή της ενέργειας και όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα. Η σύνεση πρέπει να είναι λοιπόν η γραμμή που θα ακολουθούμε. Και τώρα για το μέλλον και κυρίως για την προοπτική για το 2019 οι στόχοι και οι κύριοι κίνδυνοι που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα μας είναι έξωθεν έρχονται έξω. Δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία από πλευρά των οικονομικών ε, αναλυτών, τόσο εθνικών όσο και διεθνών, ότι ο βασικός μας στόχος, ε, η πρόκληση μάλλον, είναι η προβλεπόμενη ε, επιβράδυνση της οικονομίας της Ευρώπης και άρα και των εξαγωγών μας. Και άρα είναι πιθανόν να επιδεινωθεί το ισοζύγιο Ελπίζουμε πως αυτή η κίνηση, θα αυτή μάλλον η ύφεση θα αντικατασταθεί από την εσωτερική ζήτηση και για τη χώρα μας και για ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να επαγρυπνούμε όσον αφορά τις διεθνείς εξελίξεις. Η Ισπανία είναι όλο ένα και πιο ανοιχτή χώρα, με όλο ένα και περισσότερες διεθνείς ε, εταιρείε και άρα επηρεάζεται από το τι συμβαίνει διεθνώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Βλέπουμε πως ε, οι πρόσφατες προβλέψεις του Δέλτα Νιτάφ προβλέπουν για την Ισπανία ότι είναι μία από τις λίγες χώρες όπου δεν θα επιβραδυνθεί η ανάπτυξη. Δυστυχώς οι άλλες έχουν μία επιδείνωση της κατάστασης ε, μπροστά τους. Λοιπόν, τώρα τον λόγο έχει η κυρία Πρεβάν Σπερές για τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ πολύ χαιρόμαστε που σας βλέπουμε εδώ σε αυτόν τον οικονομικό διάλογο. Και δεν θα σας ε, εκπλήξει που θα σας ρωτήσω για τον προπολογισμό της Ευρωζώνης. Προηγουμένως όμως, θέλω να σας υπενθυμίσω κάτι. Την επιτυχία των 27 στην περίπτωση του Brexit. Νομίζω ότι δεν το τονίζουμε αρκετά. Μίλησαν με μία φωνή 27, με την κοινοτική μέθοδο και αυτό αποτέλεσε επιτυχία τελικά. Κατέληξε σε επιτυχία. Όταν υπάρχουν λοιπόν διαφωνίες, εντάσει μεταξύ των χωρών μελών, η κοινοτική μέθοδος είναι νομίζω η αριστεία και όχι μόνο για θέματα εσωτερικής αγοράς. Οπότε λυπούμε κατά κάποιο τρόπο που η διάσκεψη της Ευρωζώνης απομακρύθηκε από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ήταν ε, βέβαια μια εντάξει, μετριοπαθής πρόταση, αλλά τουλάχιστον υπήρχε και επιπλέον αναφέρονταν στο βασικό πυλώνα της Ευρωζώνης. Γιατί εξαιτία των συζητήσεων που γίνονται μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, τρία θέματα μπαίνουν στη συζήτηση. Η ανταγωνιστικότητα, που δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα ειδικό για την Ευρωζώνη. Το δεύτερο είναι η σύγκληση, που είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε συνέχεια γιατί ουσιαστικά εννοούμε αρθρωτικέ μεταρρυθμίσεις, χωρίς να μιλάμε για τις ε, ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ χωρών ελληματικών και χωρών πλεονοσματικών. Και η αναγκαιότητα για έναν προπολογισμό θα μπορούσε να αποτελέσει ε, τον παράγοντα σταθερότητας. Αυτό ήταν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ξέρετε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον Ράινερ Μπέγκαρτ έχουμε μία πρόταση η οποία χτίζει πάνω στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την εμπλουτίζει με μία άλλη λειτουργία σταθερότητας, δηλαδή με μία αποζημίωση ανεργίας ακριβώς να επίδομα ενέργεια ακριβώς για να μην ε, πλήττονται όμως τα εθνικά συστήματα, το κρατάμε χωριστά. Αυτή η συζήτηση λοιπόν ε, γίνεται. Τα συμπεράσματα για την Ευρωζώνη δεν είναι πολύ θετικά, οπότε θα ήταν σοφό να επιστρέψουμε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμπλουτίζοντας την βέβαια με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι λέτε. Απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπερές. Συμφωνώ μαζί σας βέβαια για τη σημασία που έχει να μιλάμε με μια φωνή και να έχουμε κοινό στόχο, μια κοινή φιλοδοξία για το τι θέλουμε να πετύχουμε και πού θέλουμε να βρισκόμαστε σε 5-10 χρόνια. Όσον αφορά τις συζητήσεις για την Ευρωζώνη. Πράγματι, χτες στο Eurogroup συζητήσαμε πολύ πώς να ερμηνεύσουμε τα συμπεράσματα της διάσκεψης του Δεκεμβρίου και ποιο είναι το περιθώριο ε, πάνω στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε για το 2019. Και εδώ η ερμηνεία μας είναι και αναφέρονται κατά λέξη τα συμπεράσματα της διάσκεψης, είναι λοιπόν ότι οι επικεφαλής έχουν συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία του συμπεράσματος του Δεκεμβρίου Eurogroup και COFIN συμπεριλαμβανομένης και της τεχνικής δουλειάς που πρέπει να γίνει για τη σταθεροποίηση. Τα συμπεράσματα επίσης λένε ότι πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε ένα εργαλείο συντονισμού και ανταγωνιστικότητας βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψουμε πάνω στον μεταρρυθμιστικό μηχανισμό. Άλλοι, όπως η Ισπανία, θεωρούν ότι πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ε, Σταθεροποίησεων και Επενδύσεων. Πρόκειται λοιπόν για διαφορετικές προτάσεις που βρίσκονται τώρα πάνω στο τραπέζι στα πλαίσια του μελλοντικού πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Χτες λοιπόν συμφωνήσαμε ότι θα δουλέψουμε πάνω και στις δύο βάσεις. Να δούμε πώς θα μπορέσουμε παράλληλα να προχωρήσουμε και να δούμε αυτή η λειτουργία σταθεροποίησης και προστασίας από την ανεργία πώς θα παραμείνουν στο τραπέζι. Και τελειώνω κύριε Γκολτιέρη με το εξή. Ξέρουμε ότι, και το ξέρετε πολύ καλά εσείς εδώ, ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν φτιάχνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Σιγά σιγά, ακόμα και οι ιδρυτές πατέρες το είπαν ότι δεν θα γίνει σε μια μέρα η Ευρώπη. Πρέπει να παραμείνουμε κοντά στον πολίτη, οικοδομώντας την Ευρώπη. Και όσον αφορά την ΟΝΕ, αυτό το οποίο εγώ ελπίζω και γι' αυτό δουλεύω, είναι να μην περιμένουμε την επόμενη κρίση για να έχουμε πρόοδο. Όχι, να υποφεληθούμε από την τωρινή συγκυρία που έχουμε θετική ανάπτυξη σε όλη την ε, Ευρώπη για να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, να είμαστε έτοιμοι και να μην υποφέρουμε όταν μας έρθει η επόμενη κρίση το ίδιο πολύ όπως υποφέραμε με αυτήν που μόλις τελείωσε. Πρόεδρος, ε, νομίζω ότι πολύ συμφωνούμε μαζί σας για τη λειτουργία αυτή τη σταθεροποιητική που λέμε ότι είναι κάτι αναγκαίο για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα μέσα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Άλντε, Ραμόν Τρεμόσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Γουαλτιέρη. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε εδώ. Θέλω να σας ρωτήσω για τα MPL, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 21 Νοεμβρίου του 2017 ο Μάριο Ντράγκη εδώ σε αυτή την αίθουσα, σε αυτή την ίδια κοινοβουλευτική επιτροπή ήρθε και συζητήσαμε τις αιτίε πολλές και διάφορες που οδήγησαν στα μη ξεπηρετούμενα δάνεια. Και αυτό που αποκάλεσε κύρια αιτία είπε ότι ήταν η μη τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων. Αυτή μια τήρηση ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη και στη Νότια Ευρώπη και τις ξέρουμε τις διάφορες διαδικασίες που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε βάρος πολλών χωρών που δεν έχουν ενσωματώσει τους κανόνες ε, στη νομοθεσία τους. Όμως εδώ κατηγοριούνται και πολυεθνικές και χώρες που δεν έχουν πληρώσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις διάφορες χώρες για χρόνια και έτσι έχουν ε, αναγκάσει πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κλείσουν γιατί δεν μπόρεσαν να εισπράξουν τα χρήματα που τους χρώσταγε το κράτος. Υπάρχει ένα βίντεο κάπου ένα λεπτό στο οποίο ο πρόεδρος Δράκη τα λέει όλα αυτά. Τώρα για συγκεκριμένα την περίπτωση της Ισπανίας και της πληρωμές ακόμα δεν έχει εγκριθεί ο νόμος για τις ε, κυρώσεις κατά εκείνων που δεν πληρώνουν έγκαιρα πρέπει να υπάρχουν κυρώσει. Αλλιώ, τώρα μπορεί να διευθετήσουμε αυτό το ζήτημα, αλλά σε μια επόμενη κρίση, και αν είναι μεγάλη όπως αυτή του 17, πάλι με τις καθυστερήσεις αυτές πληρωμών θα καταλήξουμε ε, στο ίδιο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε σε Τρία πράγματα έχω να πω γι' αυτό και ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Πρώτον, όσον αφορά την αιτία των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Είναι αλήθεια ότι η καθυστέρηση πληρωμών έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Στην περίπτωση της Ισπανίας, δυστυχώς, ήταν περισσότερο η φούσκα ακινήτων που οδήγησε σε τόσο κακούς ισολογισμούς στις τράπεζες και αναγκαστήκαμε να πάρουμε μέτρα, ειδικά μέτρα, ε, διαφορετικά από άλλες χώρες για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα των ε, πιστώσεων που είχαν ε, δοθεί στα πλαίσια αυτής της φούσκας ακινήτων και μέσα στην οικονομική κρίση φυσικά κανένας δεν μπορούσε να πληρώσει τα δανειά του. Τώρα τα νέα είναι αρκετά θετικά σήμερα. Οι ισπανικές τράπεζες ε, μετά από μια σημαντική προσπάθεια εξυγίανσης έχουν επίπεδα πολύ χαμηλότερα για εξυπηρετούμενα δάνεια, πολύ λιγότερο από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συζητήσαμε αυτό στο ΕΚΟΦΗΝ. Και βελτιώθηκε λοιπόν πάρα πολύ η εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών. Και ένα δεύτερο στοιχείο πολύ σημαντικό είναι ότι η Ισπανία σε αυτό το στάδιο ανάπτυξη που βρίσκεται προχωράει πιο ισορροπημένα να αντιμετωπίζει τον οικοδομικό τομέα. Υπάρχει κάποια πάλι ανάπτυξη, αλλά πιο περιορισμένη. Και βέβαια η απασχόληση που απορροφιέται από αυτόν τον τομέα, η μείωση της ανεργίας δηλαδή, εξαιτία αυτού του τομέα δεν είναι όπω ήταν παλιότερα τόσο μεγάλη. Τώρα κάτι άλλο που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι οι δημόσιε δικήσεις που πρέπει να πληρώνουν έγκαιρα, πράγματι. Για να υπάρχει η αυτονομία, τα γνωρίζετε πολύ καλά και από τη δικιά σας αυτόνομη περιφέρεια η οποία έχει πρόσβαση σε αυτούς τους μηχανισμούς χρηματοδότησης που την επιτρέπει να υποφεληθεί από την καλή κατάσταση που βρίσκεται το κράτος της Ισπανίας. Όντως, η Ισπανία πληρώνει τις αυτόνομες περιφέρειες και εκείνες με τη σειρά του μπορούν να πληρώσουν για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις που ήταν ένα πολύ βασικό στοιχείο. Και όντως, η καθυστέρηση πληρωμών ή μάλλον η μη καθυστέρηση πληρωμών από την πλευρά των περιφερειών σημαίνει ότι γίνονται και πιο αυτόνομες πράγματι. Τώρα κατά τα συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να δούμε πώς θα μειωθούν αυτές οι καθυστερήσεις πληρωμών. Με κυρώσεις. Εγώ θα ήθελα όμως να σκεφτώ και κίνητρα ή άλλα στοιχεία, τόσο πάντων πιο θετικά, τα οποία να μας επιτρέπουν να συνεχίζει η μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα πλαίσια μιας οικονομικής ανάπτυξης που μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη όσο θα θέλαμε και που περιορίζει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να πληρώσουν αμέσω. Ευχαριστώ. Ουρτασούν εκ μέρους των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ Υπουργέ. Καλώς ορίσατε στην ε, απόψινή συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών και εγώ εμένα μου άρεσε αυτό το backstop for the people που, αναφέ, που είπατε εσείς ως ε, έκφραση αλλά ε, ιδιαίτερα όσον αφορά το, το το τι συνέβη, συμβαίνει ε, με, τα σπίτια και συμβαίνει σε πολλές πόλεις στην Ευρώπη. Η δυνατότητα δηλαδή ρύθμισης των ε, νοικίων. Υπάρχει στη Γερμανία ας πούμε ε, ένα σύστημα που βασικά με βάση συγκεκριμένες τιμές μπορεί κανείς ε, είτε να επιβάλλει ε, πρόστιμα στα σπίτια που νοικιάζονται πολύ πάνω από αυτές τις τιμές είτε να προωθήσει τα σπίτια που νοικιάζονται πολύ χαμηλότερα από αυτές τις τιμές ε, εν πάση περιπτώσει βάζει ανώτατα όρια για συγκεκριμένες ζώνες, για συγκεκριμένες περιοχές γι' αυτό δεν υπάρχει και μαύρη αγορά υπάρχει και ένα πρόγραμμα στη Γαλλία τώρα που ονομάζεται ΕΛΑΝ μετά από από την άνοδο την αστυνομική των ηλικίων 2015 με 2017 εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί δεν μπορέσαμε εμείς να εισάγουμε αυτό το μέτρο ενώ έχουν επιτυχεί αυτά τα συστήματα στη Γαλλία ή στην ε, Γερμανία γιατί η στη γερμανια γιατι η δικη σας κυβέρνηση δεν κατάφερε να περάσει τι συνέβη στο, ε, ε, στη Βουλή Μπορούμε λοιπόν μήπως να το ξανασυζητήσουμε. Τι χρειάζεται να γίνει μήπως και περάσει ένα τέτοιο σύστημα και για την Ισπανία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ορτασίν. Δεν θέλω να φέρω εδώ στην έδρα του Ευρωκοινοβουλίου μια συζήτηση που έχει νόημα περισσότερο στην Ισπανική Βουλή. Σας ευχαριστώ ωστόσο για την ερώτησή σας γιατί το θέμα της πρόσβασης από πλευράς όλων των πολιτών σε, μια, σε ένα αξιοπρεπές ε, ε, σε μια αξιοπρεπή στέγη ήταν ε, μέρημνα της κυβέρνησής μας από την πρώτη μέρα ε, και είχα την ευκαιρία σε διάφορα πλαίσια να εξηγήσω την θέση μας. Καταρχάς όσον αφορά την πρόσβαση στη στέγη σαν ακίνητη περιουσία. Φτάσαμε σε, με μεγάλη καθυστέρηση της μεταγραφής των οδηγιών, των ευρωπαϊκών οδηγιών στην Ισπανία, όπως ας πούμε πούμε, για παράδειγμα με, την, με την οδηγία για τα ενυπόθηκα δάνεια. Φτάσαμε με την επιτεχημένη ε, διαδικασία στο Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να έχουμε μια τέτοια νομοθεσία που να ε, προστατεύει τους πολίτες. Ε, μέσα από την κοινοβουλευτική του πορεία αυτός ο νόμος μπορεί όντως να στηρίξει τα πιο ευάλωτα άτομα που προσπαθούν προσπαθούμε να θεσπίσουμε διάφορες ρήτρες ασφαλείας πριν να φτάσουμε σε κατάσταση έξωσης και να θέσουμε όρους οικονομικούς όσο γίνεται πιο δίκαιους για να μπορούμε να προστατεύσουμε τους πολίτες. Πολύ σημαντικό αυτό για μια χώρα όπως η δική μας, όπου ο περισσότερος κόσμος έχει στην ιδιοκτησία του ε, ένα σπίτι. Αλλά πρέπει όντω να μιλήσουμε για το θέμα των ε, ενοικίων που δεν μπορούμε με ένα μαγικό ραβδί να το ρυθμίσουμε. Αυτό που είδαμε στη χώρα μας τελευταία χρόνια ήταν ότι σταδιακά μειώθηκε η προσφορά ε, ενοικιαζόμενων ε, διαμερισμάτων ε, κοινωνικού τύπου, δημόσια δηλαδή ε, καταλήματα. Αυτή είναι η κατάσταση. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εργάζεται πάνω σε αυτό. Πρέπει να έχουμε και ένα συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε με το νομοσχέδιο στο οποίο αναφέρομαι και ε, προσπαθούμε να θεσπίσουμε και έναν μηχανισμό κοινωνικού τύπου ώστε να αποφεύγεται η έξωση σε περιπτώσεις όπου είναι πιο ευαίσθητες. Όσον αφορά το νομοθετικό διάταγμα, Έχουμε βάλει συγκεκριμένε ε, τάξεις για να αποφεύγονται οι εξώσει. Επίσης έχουμε θέσει όρια στα τουριστικά καταλήματα. Ε, μια διαδικασία που είναι πολύ γνωστή και σε άλλες χώρες, σε άλλες μάλλον ευρωπαϊκές πόλεις. Ε, και προσπαθούμε επίσης να θεσπίσουμε μέτρα ε, για να μπορούμε να ελέγχουμε ε, τι γίνεται με τα σπίτια που νοικιάζονται στα πιο χαμηλά νίκια, δηλαδή γύρω στα 600 ευρώ, δηλαδή οι πιο ευάλωτες ομάδες. Γι' αυτό ε, και έτσι προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τις πιο επίγουσες πτυχές, αυτό δηλαδή που μας ζητήθηκε από την κοινωνία και λυπούμε που δυστυχώ δεν είχαμε την απαραίτητη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο για να υιοθετήσουμε αυτά τα επίγοντα μέτρα που δεν είναι εμπόδιο Χρειάζεται ίσως να οριμάσουν περισσότερο ή κάποια άλλη νομική βάση. Είναι ενδιαφέρον, ε, ενδιαφέρουσες οι εμπειρίε που εσείς αναφέρατε. Οι εκθέσεις που εγώ μπόρεσα να διαβάσω ίσως να μην είναι τόσο αισιάδεξες ή τόσο θετικές σε σχέση με τον αντίκτυπο που είχαν αυτά τα μέτρα στις ε, τιμές των ενοικίων, αλλά σίγουρα οι διεθνείς προσπάθειες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως έμπνευση για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά στην χώρα μας, όπως γίνεται και αλλού. Ευχαριστώ, Μιγγέλ Ούρμπαν Κρέσπο, Γκουε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ. Θα συνεχίσω με το θέμα που άνοιξε ο συνάδελφος Σουρτασούν. Γιατί δέκα χρόνια μετά την κρίση βρισκόμαστε πάλι μπροστά σε μία φούσκα ακινήτων που τροφοδοτείται πολιτικά για να σωθούν οι τράπεζες, οι ισπανικές τράπεζες. Όπως ξέρετε, ε, το ότι μπήκανε ποσά στην ισπανική αγορά αυτό ήταν μια κοινωνική καταστροφή για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που εξακολουθούν να είναι θύματα μιας ε, φούσκας ακινήτων με ένα σωρό καταχρήσεις που γίνονται σε βάρος των ε, οικογενειών αυξάνοντας ε, τα ενίκια και αναγκάζοντας έτσι τις οικογένειες να φύγουν από τα σπίτια τους. Έχουν καταγγελθεί οι πρακτικές αυτές στην Ισπανία ε, το κυπερημερίας για παράδειγμα. Όμως δεν εκβιάζονται εδώ πέρα μόνο οι οικογένειες, εκβιάζεται και η ίδια η κυβέρνηση η οποία απειλείται γιατί λένε ότι θα σταματήσουν οι εταιρείε αυτές τις επενδύσεις τους αν δεν υπάρχει αύξηση στα ενίκια. Να ρωτήσω κάτι λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Πιστεύετε ότι μια αγορά όπως αυτή των ακινήτων δεν πιστεύετε ότι χρειάζεται ρύθμιση στις τιμές για να μπορέσει να έχει και μια κοινωνική λειτουργία. Θεωρείτε ότι οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ώστε να δίνουν... ώστε να μεταφέρονται τα δάνεια κακής ποιότητας θα μπορούσε να ήταν μια λύση για εκατοντάδες οικογένειες. Και τι πιστεύετε για την Ευρωπαϊκή Οδηγία για αυτούς που αγοράζουν ε, τα δάνεια και που τελικά τα μεταφέρουν σε ολόκληρη την Ευρώπη και φέρνουν φρέσκο χρήμα στην αγορά κινήτων. Δεν θα έπρεπε να διευρυνθεί η κοινωνική κατοικία. Δεν θα έπρεπε να ενισχυθεί μια τέτοια κοινωνική κατοικία με ενίκια τα οποία να μπορεί να πληρώσει ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ουρμπάν. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για αυτό το θέμα, θα σας απαντήσω κάπως συνοπτικά. Πρώτα απ' όλα ζήτησα από τον συνάδελφο να μου βρει κάποια στοιχεία, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάει κανείς για φούσκα κινήτων πάλι. Όχι. Οι τιμές στο κέντρο κάποιων πόλεων μπορεί να είναι πολύ ψηλές, αλλά δεν συγκρίνεται με αυτό που είχαμε παλιότερα. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε σήμερα για νέα φούσκα κινήτων. Ω Υπουργό ε, Οικονομικών καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να αφήσω να ε, κυκλοφορεί εδώ ένα τέτοιο μήνυμα που δεν είναι σωστό. Δεύτερον, συμφωνώ με την ανησυχία σας και τη συμμερίζομαι για το ότι δεν καταφέραμε να προστατεύσουμε το κόσμο στο παρελθόν. Γι' αυτό και είμαι ικανοποιημένη που με τον νέο νόμο για τα στεγαστικά δάνεια μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των μηνών που δεν πληρώνει κανείς πριν ξεκινήσουν οι εξώσεις. Δεύτερον, ε, προστατεύονται ε, τα συμφέροντα των καταναλωτών όταν υπάρχουν οι τόκοι περιμερίας. Έπειτα υπάρχει ένας κώδικας διοντολογίας ώστε πριν φτάσουμε στην έξωση, αν κάποιο άτομο είναι ευάλωτο, πρέπει η τράπεζα να του προσφέρει διάφορες δυνατότητες επαναδιαπραγμάτευσης κλπ. κλπ. Η νέα αυτή νομοθεσία ακριβώς καθησυχάζει κάποιες από τις ανησυχίες που αναφέρατε εσείς. Έπειτα, η έξωση ευάλωτων ατόμων που δεν πληρώνουν ε, νίκη και δεν έχουν άλλο σπίτι, όντω είναι ένα δράμα. Είναι μια τραγική κατάσταση. Συμφωνώ και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό και η κυβέρνηση αυτό ακριβώ προσπαθεί να κάνει και με το νόμο αυτό που περιλαμβάνει υποχρέωση διαβούλευσης του δικαστή με τις κοινωνικές υπηρεσίες πριν αποφασιστεί η έξωση. Φροντίζουμε δηλαδή να προσφέρουμε κάποιες εγγύησεις ώστε να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους πολίτες. Γι' αυτό και θέλαμε αυτό το νόμο με ισχύ απευθείας. Έπειτα, μιλήσατε για εκβιασμό. Όχι, δεν εκβιάζει κανένας την Ισπανική κυβέρνηση. Κάποιοι το πέταξαν αυτό, το άκουσε ο κόσμος, αλλά δεν ισχύει. Δεν έχουν προσθέσει τίποτα. Δεν εκβιάζεται από κανέναν η Ισπανική κυβέρνηση. Τέλος, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και με αυτό ξεκίνησα όταν απάντησα στον ε, κύριο Ρτασούν πριν από λίγο. πρέπει να αντιμετωπίσουμε διάφορα μέτωπα. Ένα από αυτό είναι η προσφορά κατοικία, κοινωνική με λογικά νίκια. Αυτό προσπαθούμε να ανακτήσουμε. Γι' αυτό και από την αρχή ο Γενικό Γραμματέα ακριβώ του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι και αυτό που είναι πιο υπεύθυνο για αυτά τα θέματα, ξεκινήσαμε να το ξαναβλέπουμε αυτό με ένα σχέδιο που θέλουμε να αναζωογονήσουμε, να δούμε πού θα μπορούσαν να υπάρχουν τέτοιες κατοικίες ώστε να μπουν στην αγορά. Την προηγούμενη εβδομάδα υπέγραψα την παράταση του Συμφώνου Κοινωνικής Κατοικίας με τις αρμόδιες αρχές, ώστε 10.400 κατοικίες, αν δεν διατέθηκαν για πιο ευάλωτα άτομα και την προηγούμενη εβδομάδα υπογράψαμε και την παράταση αυτού του σχεδίου για την κοινωνική κατοικία. Και η υπόλοιπη κυβέρνηση επίσης δουλεύει για ένα σχέδιο κατοικίας ώστε να έχουμε καλές ε, συνθήκες. Οι λύσει φυσικά δεν μπορεί να είναι από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν κρατάμε το μαγικό ραβδί, αλλά από την πρώτη μέρα αρχίσαμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση στα διάφορα μέτωπα τα οποία επηρεάζουν την αγορά κατοικία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Μάρκο Τζάνι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Στην ε, εισήγησή σας ε, μιλήσατε για την πρόοδο της ισπανικής οικονομίας και για το τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνησή σα και τι θα προσπαθήσει να κάνει τους επόμενους μήνες. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις ε, που είναι όμως γενικότερες για την πρόοδο τη οικονομία ε, στην Ευρώπη. Εδώ και ένα χρόνο υπάρχουν ισχυρά μηνύματα όλο ένα και πιο έντονα για επιβράδυνση τη παγκόσμια οικονομία και κυρίω για επιβράδυνση τη ευρωπαϊκή οικονομία. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, δεν φαίνεται οι εκλογές των χρόνων της κρίσης ε, και τα σφάλματα που διπράχθησαν στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων και μάλιστα ο πρόεδρος Γίνκερ ε, ε, έκανε αρκετά ασφάλματα περνάμε προς έναν οικονομικό κύκλο προς επιβράδυνση αλλά εξακολουθεί η ευρωπαϊκή πολιτική και εσείς το είπατε σε κάποια σημεία της ομιλίας σας επιμένει στη μείωση του δημοσίου χρέου, στις πολιτικές σύνεσει σε σχέση με τον προπολογισμό που μπορεί να επιδεινώσουν την επιβράδυνση που ήδη έχει ξεκινήσει. Θέλω να καταλάβω λοιπόν κάπω τη γνώμη σα για μια ριζική αλλαγή, κυρίως ενώπιον αυτή της επιβράδυνση της οικονομίας ε, και επίσης ε, αυτή η συζήτηση που ξεκινά για το, τη σχέση χρέους ΑΕΠ ε, του 70% μήπως αυτό είναι κάπως αναχρονιστικό και έπειτα ε, το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωζώνης το οποίο έχουμε δανειστεί ε, δεν θα έπρεπε αυτό το μοντέλο να το ξαναδούμε εκ βάθρων, γιατί έτσι η οικονομία της Ευρωζώνης εξαρτάται υπερβολικά από τις αποφάσεις που δεν ε, μπορεί να ελέγξει σε μια περίοδο δηλαδή όπου οι Αμερικανοί είναι πιο προσεκτικοί και έχουν αλλάξει στάση για το θέμα των, ε, ε φόρων. Η Κίνα επίσης επιβραδύνει και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε με τον Brexit, το να στοχεύουμε μόνο στην οικονομία που εξάγει αντί να... Ε, βασιζόμαστε στην εσωτερική ζήτηση, μήπως είναι αδυναμία. Ευχαριστώ. Είναι ενδιαφέροντα τα όσα είπατε. Ποια είναι δηλαδή τα διδάγματα που κομίσαμε από την κρίση. Για την περίπτωση της Ισπανίας νομίζω πως ναι μάθαμε από την περίοδο της κρίσης. Είδαμε πως δεν είναι λογικό να πιστεύουμε ότι σε μια κατάσταση οικονομικής αστάθειας ο δημόσιος τομέας θα μπορέσει να συνεχίσει με στρατηγική Χωρί χωρίς να τιμωρηθεί από τις, οικονομικές, από τις ε, ε, χρηματοπιστωτικές αγορές. Όπως είπατε, μειώνεται ο όγκο των χρημάτων των φορολογούμενων που πρέπει να πληρώνουν ε, και να, να εξυπηρετούν το χρέος. Ε, άρα λοιπόν πρέπει να μειωθούν, ε, να μειωθούν τα επιτόκια και να συμβάλλουμε ε, στην ανάπτυξη, στην παιδεία, στην υγεία και τα λοιπά, στις κοινωνικές πολιτικές εν γέννη. Καταλάβαμε πως η οικονομική σταθερότητα είναι βασική για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το χώρο, να ασκήσουμε πολιτικές και επιπλέον το δημόσιο χρέος δεν είναι μόνο πρόβλημα ε, κρατικό είναι και θέμα δικαιοσύνης ανάμεσα στις γενιές. Δεν μπορούμε να χρεώνουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας δηλαδή. Πιστεύω λοιπόν ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι πολιτική ε, σταθερή ε, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε πιο περισσότερο φιλόδοξους στόχους ε, ε, και να μην θέτουμε σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη. Η κυβέρνησή μας μάλιστα είχε στόχο μείωση του χρέους στο 1,8% λόγω της, της, των προβλημάτων στο Βουλή και στην Γερουσία χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1,3% και ελπίζω πως θα μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε την αρνητική, τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής. Όμως μιλάμε για ε, δέκατα της μονάδας και ελπίζουμε πως θα καταφέρουμε να μειώσουμε το χρέος για τους λόγους που εσείς είπατε και όχι για ότι επειδή μας υποχρεώνουν τα κοινοτικά όργανα. Έπειτα συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι σε αυτό το σενάριο επιβραδυμένης ανάπτυξης των διεθνών αγορών, η εσωτερική ζήτηση θα πρέπει να είναι ο βασικός κινητήρας ανάπτυξης. Για την Ισπανία, τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση ήδη το Δεκέμβριο, ήδη, δηλαδή η αύξηση της αγοραστικής δύναμης των οικογενειών, η αύξηση του ελάχιστου μισθού κτλ. Νομίζουμε πως θα έχει θετικό αντίκτυπο στην κατανάλωση και ελπίζουμε πως θα παραμείνει σταθερός ο δυναμισμός επενδυτικός που διαπιστώνει διαπιστώθηκε στην Ισπανία το 2018 προς το τέλος κυρίως το δεύτερο μισό ακριβώς έτσι ώστε η εσωτερική ζήτηση να τονωθεί και η ίδια ανάλυση ισχύει και για την Ευρωζώνη. Σας ευχαριστώ. Ο Ζίκφριτ Μορεσάνα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ ξανά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαμε πολύ καλή επαφή όταν ήσασταν βουλευτή στην Επιτροπή Προπολογισμών και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό στο μονάχο. Τρει ερωτήσει. Η πρώτη σχετίζεται με τι οικονομικέ εξελίξει στην Ισπανία. Μιλήσατε για τι τελευταίε μακροοικονομικέ εξελίξει και σχετίζεται με την αύξηση του βασικού μισθού. Αποφασίσατε να τον αυξήσετε κατά 22% αρχέ του έτου. Το ερώτημά μου είναι τι ε, ε, αξιολογείς θεωρείτε ότι αυτό θα έχει όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, το χρέος και την απασχόληση, γιατί βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η ανάκαμψη και η ανάκτηση της ε, ανταγωνιστικότητας της ισπανικής οικονομίας και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τα αποτελέσματα της ε, δημοσιονομικής εξυγένσης. Δεύτερον, οι συστάσεις αναχώρα του 2017 μιλάνε για μειωμένη ικανότητα καινοτομία των ισπανικών εταιριών επειδή υπάρχει μια ασυμφωνία δεξιοτήτων και προτείνουν επενδύσεις στην εκπαίδευση. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό και τρίτη ερώτηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης. Ε, ε Γι' αυτό θέλω να σα ρωτήσω τι ποσό, τι όγκο, τι τάξη μεγέθου θεωρείται ρεαλιστικό δεδομένου του ότι θα πρέπει και να αυξηθεί ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι σχέση βλέπετε μεταξύ των χωρών τη Ευρωζώνη και των μη κρατών μελών τη Ευρωζώνη. γιατί βεβαίω αυτό θα αφορά κυρίω την Ευρωζώνη αλλά θα χρηματοδοτείται από τον κοινοτικό προπολογισμό στον οποίο συνεισφέρουν όλα τα κράτη-μέλη. Τι άποψη έχετε από αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μουρεσάν. Χαίρομαι που σας ε, ξαναβλέπω. Δεν θυμόμουν ότι ήσασταν και στην Επιτροπή αυτή. Τρία... Τρεις απαντήσεις στις τρεις ερωτήσεις σας για τον ε, βασικό μισθό. Ε, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να κλείνουμε τα κενά. Δηλαδή, ο βασικός ο λόγος βασικού μισθού με μέσο μισθό στην Ισπανία ήταν σαφώς κάτω από τις υπόλοιπες ε, χώρες του ΟΣΑ και είχαμε σοβαρή μείωση ε, τα τελευταία χρόνια, οπότε έπρεπε να γίνει μια ξεκάθαρη ελεγγύη για να ανακτήσουμε έναν κατάλληλο βασικό μισθό, ειδικά σε μια χώρα όπου είδαμε τα τελευταία χρόνια την εμφάνιση φτωχών εργαζομένων, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και δεν τα καταφέρνουν στο τέλος του μήνα. Δεν τα βγάζουν πέρα. Επίσης είναι σημαντικό από την ε, σκοπιά της ισότητας των φύλων. 70% των ατόμων που εργάζονται με το βασικό μισθό στην Ισπανία είναι γυναίκες, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να κλείσει το μισθολογικό χάσμα. Τρίτον, έχουμε τα στοιχεία, εντάξει τα μοντέλα διαφέρουν όσον αφορά τα συμπεράσματα, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι ε, τις χρονιές που είχαμε αύξηση του βασικού μισθού δεν είχαμε κάποια μείωση της απασχόλησης. Αντιθέτως, είχαμε αύξηση της απασχόλησης, ειδικά της νεολαίας, που ε, υποτίθεται ότι θα επηρεαζόταν περισσότερο. Και η τελευταία ένδειξη που έχουμε είναι ότι τον Δεκέμβριο, που ήταν ήδη γνωστή η αύξηση του βασικού μισθού, τα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας ήταν ιδιαίτερο θετικά, δηλαδή δεν σταμάτησαν οι προσλήψεις. Βεβαίως πρέπει να τα παρακολουθούμε αυτά στενά, όπως είπατε. Δεύτερον, για αυτή την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μου και σε πολλές χώρες ε, στην Ευρώπη. Και θέλουμε πραγματικά να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, στο ανθρώπινο κεφάλαιο και να ευθυγραμμιστούν αυτά με τις ανάγκες ε, των επιχειρήσεων. Και ακριβώς θα δούμε όλο αυτό το θέμα του προφίλ για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για να μπορέσουμε δηλαδή να προσαρμοστούμε στις ανάγκες της νέας οικονομίας, ειδικά την επανάσταση που βλέπουμε στα ψηφιακά ζητήματα. Και τέλος, αυτή είναι η ερώτηση στην οποία μάλλον δεν θα απαντήσω, γιατί ξέρετε, επειδή ήμουν και στην Επιτροπή που κάναμε την πρόταση, γνωρίζετε το δημοσιονομικό περιθώριο που υπήρχε τότε. Τώρα που προσωπώ την Ισπανία βεβαίως ίσως έχω διαφορετική άποψη, αλλά επιφυλάσσομαι μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αλλά οι συγκητές του Κοινοβουλίου μας είναι νομίζω επαρκώς φιλόδοξοι, αλλά ρεαλιστές, ελπίζω. Χώνας Φερνάντες. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας για να μάθουμε από πρώτο χέρι το πρόγραμμα της ε, χώρας μας, αλλά και τις προοπτικές που βλέπει η Ισπανική κυβέρνηση στα πλαίσια της Ευρώπης. Σχόλια πρώτα. Για την σημαντική καθυστέρηση της κυβέρνησης προκειμένου να ενσωματώσει την οδηγία για τις υποθήκες. Αλλά θέλω να μου πείτε τι γίνεται με τη σημερινή συζήτηση μετά την πρότασή σας για να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός μακροεποπτικός, όπως επίσης και για τα μακροεποπτικά μέσα για να διευκολυνθεί η Τράπεζα της Ισπανίας, η διαδικασία διαπραγματεύσεων ήταν δύσκολη από ό,τι φαίνεται. Και το Λαϊκό Κόμμα βλέπει δυσκολίες και μπορεί να μην συμφωνήσει. Εσείς τι λέτε. Δεύτερον, για την συζήτηση που γίνεται επιμονή μου βάσεως όσον αφορά τον διακυβερνητικό και τον κοινοτικό μηχανισμό. Εσείς αναφερθήκατε στην ε, αλλαγή του μηχανισμού σταθερότητας. Υπάρχει η συνθήκη η κυβέρνηση εκτός από ευρωπαϊστική που δηλώνει ότι είναι θα χρησιμοποιήσει την κοινοτική μέθοδο αλλά θα διατηρήσει και τον έλεγχο. Και τρίτη μου ερώτηση έχει να κάνει με την μεταρρύθμιση της Νομισματικής Ένωσης, με το ΕΝΤΙΣ και με τον προπολογισμό. Για τον προϋπολογισμό λίγα έχω να πω όντω πρέπει να έχει μια λειτουργία σταθεροποίηση, το είπατε κι εσεί. Αλλά θέλω να μου πείτε τη διαδικασία διαπραγματεύσεων για το ΕΝΤΙΣ. Πώ τη βλέπετε, Πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε του επόμενου μήνε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Φερνάντες. Τρία σημαντικά θέματα. Για την καθυστέρηση της οδηγίας. Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, είχα 12 κοινοτικέ οδηγίες. Κάποιες ήταν σε κρεμότητα εδώ και χρόνια και δεν είχαν ενσωματωθεί στην νομοθεσία. Δεν ξέρω γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δεν θέλησε να τις προχωρήσει, να τις πάει στο Κογκρέσο. Πάντως, σαν προτεραιότητα εμείς θέσαμε να ενσωματωθούν στην νομοθεσία. Και παρά την ε, κατάσταση στη Βουλή ξέρετε ότι έχουν πολύ περιορισμένη πλειοψηφία, δεν έχουμε καν, καταφέραμε παρόλα αυτά να περάσουμε εννέα οδηγίε. Βέβαια η διαδικασία καταλαβαίνετε ότι δεν τελειώνει ποτέ, γιατί όσο ενσωματώνεις μια οδηγία, τόσο εμφανίζονται καινούργιε που πρέπει να ενσωματώσεις. Έγιναν όμως πολλά πράγματα αυτούς τους 7 μήνες και απομακρυνόμαστε από μια κατάσταση που είχαμε ακόμα και απειλές για κυρώσεις όπου θα αναγκαζόμασταν να πληρώνουμε εκατομμύρια μη ενσωματώνοντας τις οδηγίες στην Ομοθέσια μας. Τώρα για τα εποπτικά την ε, Τράπεζα της Ισπανίας, ε, ασφαλής κλπ. Υπάρχουν ε, όντως νέα εργαλεία μακροεποπτικά. Για κάποια τα ξέραμε. Κάποια άλλα τα εφαρμόζουμε για πρώτη φορά, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε εν δυνάμει φούσκες, όχι μόνο στο στεγαστικό τομέα, αλλά και στα χρηματοδοτικά μέσα. Κάποιοι δεν κατάλαβαν ότι πήγε το θέμα. Όπως λέγαμε και πριν, οι μεταρρυθμίσεις είναι καλό να γίνονται όταν τα πράγματα πάνε καλά. Μην περιμένουμε την επόμενη κρίση. Και τώρα λοιπόν αυτό θα έπρεπε να γίνει για τις ε, μακροεποπτικές μεταρρυθμίσεις. Τώρα που έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας και όχι την τελευταία στιγμή βλέποντας ότι φτάσαμε σε κρίση. Εγώ ήξερα ότι είχαμε ήδη εγκρίνει, αλλά ναι, σωστά, έχει δίκιο ο, ο συνάδελφος, ακόμα δεν έχουν περάσει. Η Ισπανία πάντως με την Ιταλία είμαστε οι τελευταίες χώρες για τη μακροποπτική αρχή, το οποίο είναι περίεργο, γιατί ακριβώς ένας από τους λόγους που μας οδήγησε στην οικονομική κρίση πριν από 10 χρόνια είναι ότι δεν υπήρχε συνολική εποπτική εικόνα. Η Ισπανία πάντως είναι υπέρ της κοινοτικής μεθόδου η αποστολή, ο προορισμός τελικά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ε, πρέπει να είναι ακριβώς αυτό. Και η Ισπανική κυβέρνηση θέλει να περάσουμε σε κάποια θέματα από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει, να θέλουμε να είμαστε πραγματικά φιλόδοξοι όσον αφορά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Τέλο, για την εγγύηση καταθέσεων. Το έντυση είναι ένα λεπτό ζήτημα αυτό. Το γνωρίζετε πολύ καλά εσεί. Γιατί στι διάφορε χώρε υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα και διαφορετικέ ευαισθησίε. Και πολύ έντονε, μάλιστα, όσον αφορά την εγγύηση καταθέσεων. Πιστεύω ότι το ότι έχουμε σαν στόχο να καταλήξουμε τον Ιούνιο σε κάτι αυτό βοηθάει. Εμείς προτείναμε για να ξεμπλοκάρει η κατάσταση, η οποία εδώ και πολύ καιρό στο Συμβούλιο παραμένει μπλοκαρισμένη, καλό θα ήταν να αλλάξουμε κάπως ε, το παιχνίδι και να φωνάξουμε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ε, να μας πούν Δυστυχώ δεν καταλήξαμε σε αυτή τη συμφωνία. Αλλά εγώ θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρξει πρόοδος. Και αν μη τι άλλο θα υπάρξει πολιτική συζήτηση τον Ιούνιο από τους ε, επικεφαλείς. Και να μπορέσουμε έτσι να συνεισφέρουμε και εμείς ως Ισπανία και βασιζόμενοι στην εμπειρία που συλλέξαμε τα 17 χρόνια. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Σα ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Θα ήθελα να αναφέρω ένα θέμα το οποίο ανέφερε ο κύριος Μάτο. Ο, η τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και ανάπτυξη είναι βασική πρόκληση όσον αφορά τις οικονομίες της Ένωσης που θέλουν να είναι δίκες και ε, ισότιμες. Επίσης, ε, ε, Γι' αυτό δεν θα πρέπει οι δημόσιες πολιτικές ε, να παραβαίνουν τη δημοσιονομική πειθαρχία και ισορροπία, ωστόσο να μπορούν να μειώνουν το χρέος. Ωστόσο φαίνεται να αμφισβητείται αυτή τη στιγμή η πορεία της Ισπανίας ενώπιον ενό σενάριου σημαντικής αύξησης των δημοσίων δαπανών όπως προβλέπει το σχέδιο προπολογισμού σας οι συμπεριφορές της ε, οικονομικής ανάπτυξης όπως και του δημόσιου χρέους σύμφωνα με την τελευταία ε, ε, μελέτη της Κομισιόν είναι αντίθετη ε, με ένα πιο περιορισμένο δημόσιο χρέος. Ποιο είναι, λοιπόν, ποιος είναι λοιπόν ο στόχος σας κύριε Υπουργέ όσον αφορά το έλλειμμα του προϋπολογισμού για τα επόμενα ε, χρόνια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κερόλτο. Όπως προσπάθησα να εξηγήσω, η δέσμευση της ε, κυβέρνησης της Ισπανίας σε σχέση με το δημοσιονομική πειθαρχία εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό μας από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων. Είναι προφανές πως η Ισπανία πρέπει να συνεχίσει σε αυτή την πορεία που θα μας επιτρέψει να μειώσουμε το βάρος του δημόσιου χρέους όπως σας είπα και πριν από λίγο. Και αυτό εξηγεί γιατί προτείναμε ένα σχέδιο προπολογισμού το οποίο έχει πολύ φιλόδοξο στόχο μείωση ε, του ελλείμματος 2,8 με 1,3 ε, μάλλον από το 2,8 στο 1,3 του ΑΕΠ μέσα στο 2019. Αυτό είναι ο γεγονός. Είναι η πιο σημαντική, πιο φιλόδοξη μείωση από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας ακολουθεί η Φιλανδία και η Ισπανία θα έχει το πιο φιλόδοξο στόχο μείωσης του χρέους. Αν με ζητάτε ακόμη περισσότερη φιλοδοξία, δεν ξέρω μέχρι που θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Το σχέδιό μας ε, κυρίως στοχεύει την αύξηση των εσόδων. Γιατί? Διότι ο μέσος όρος δημόσιων δαπανών σε σχέση με το ΑΕΠ στην Ισπανία είναι πολύ κάτω από τον κοινοτικό. Δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο για μείωση των δημοσίων δαπανών, κυρίως όταν έχουμε 70% δαπανών σε σχέση με κοινωνικές πολιτικές, παιδεία, υγεία και κοινωνικές πολιτικές. Όμω το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο είπε ότι το περιθώριο ελιγμού για τη μείωση των δημοσίων δαπανών δεν είναι πολύ μεγάλο και γι' αυτό και οι συστάσει προς τη χώρα μας στόχο είχαν την αύξηση των εσόδων. Και επίσης επειδή τα ποσοστά εσόδων σε σχέση με το ΕΠ είναι πολύ κάτω από τον μέσο, κοινοτικό μέσο όρο, είμαστε στο 38% ενώ η υπόλοιπη ένωση μέσω όρος είναι 45% για να μην μιλήσουμε για τις σκανδιναβικές χώρες που είναι οι πιο φιλόδοξες όσον αφορά τα έσοδα, τα δημόσια έσοδα. Γι' αυτό και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την καλή οικονομική κατάσταση για να θεσπίσουμε μια βάση, ε, πιο στέρεα βάση εσόδων, ώστε το χρέος να μην επιδεινωθεί μόλις θα υπάρξει επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, πράγμα που ελπίζω θα γίνει όσο γίνεται αργότερα. Γι' αυτό η στρατηγική μας θεωρούμε πως είναι η πιο υπεύθυνη, να προσπαθήσουμε να κάνουμε δηλαδή μια διαθετική προσαρμογή για να έχουμε μια πιο υγιή σελίδα για το δημόσιο τομέα και να προσεγγίσουμε την Ισπανία στο κοινοτικό μεσόωρο όσον αφορά τα έσοδα, ε, ε, το φόρο επί των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και τον ψηφιακό φόρο, ψηφιακό φόρο που τα έχουμε ήδη συζητήσει Αυτοί οι φορείς ε, μέχρι τώρα είχαν περισσότερα πλεονεκτήματα, ήταν πιο ευνόμενοι από ότι οι παραδοσιακοί φορεί. Ευχαριστώ. Κύριο Σάντζ. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, οι προοπτικέ ανάπτυξη για ολόκληρη την Ευρωζώνη πέφτουν και έχουμε και τι ανησυχίε που προκαλεί το Brexit. Εν τω μεταξύ, τα επίπεδα των επενδύσεων είναι μειωμένα, ειδικά των δημοσίων επενδύσεων ενώ έχουν δημιουργηθεί θέσεις εργασίας, αλλά οι συνθήκες δεν είναι πολύ ικανοποιητικέ. Υπάρχει μια γενική αίσθηση ότι δεν έχει βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο, ειδικά για τα χαμηλότερα εισοδήματα. Δεν θεωρείται ότι έχει φτάσει η στιγμή να κάνουμε κάποια πρωτότυπη σκέψη ε, όταν βλέπουμε ακριβώς το πώς εξελίσσονται οι κανόνες ε, της Ευρωζώνης. Εντάξει, μπορούμε να έχουμε οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αλλά αυτό οδηγεί σε κοινωνική αστάθεια. Κάποιοι λένε ότι κάπου στη μετάφραση έχουν χαθεί οι ιδέες της κοινωνικής Ευρώπης. Οι κανόνες της Ευρωζώνης μήπως φρενάρουν τις δημόσιες επενδύσεις, ειδικά όταν οι κυβερνήσεις ε, πρέπει να δώσουν κάποιες απαντήσεις στις προσδοκίε των ανθρώπων για καλύτερες συνθήκες. Αντί οι κυβερνήσεις να κάνουν παραχωρήσεις ε, κοινωνικών επιδομάτων λόγω ταραχών ή επειδή έρχονται δύσκολες εκλογές. Μήπως θα μπορούσε η Ευρωζώνη να συντονίσει μια κοινωνική απάντηση. Παραδείγματο χάρη να αντιγράψει αυτό το οποίο έκανε η βρεζονη να συντονισει μια κοινωνικη απαντηση παραδειγματο χαρη να αντιγραψει αυτο το οποιο εκανε η ισπανια και να υπάρξει ένας συντονισμός για μια αύξηση 5% του βασικού μισθού ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, θεωρείτε ότι είναι λογικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ιδέες σας ε, και για το ότι ζητάτε πρωτοτυπία. Αυτό ακριβώς ε, προσπαθούμε να κάνουμε ε, η νέα κυβέρνηση από την πρώτη μέρα και ακριβώς προσπαθήσαμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ δημοσιονομικής αρχίας και κοινωνικών πολιτικών. Συμφωνώ πλήρως οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, πρέπει να θεωρούν ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και οι εθνικές αρχές ενδιαφέρονται για αυτούς. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους εχνοκράτες ή τις τράπεζες, ε, πρέπει να αφορά όλους τους ε, πολίτες. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να βρούμε την σωστή ισορροπία. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να βρούμε την σωστή ισορροπία, όπως είπαμε, και των δημοσίων επενδύσεων και μια δημοσιονομική πολιτική η οποία θα είναι προληπτική, αξιόπιστη και στο μέτρο του δυνατού συντονισμένη ειδικά εντός της Ευρωζώνης. Γιατί όσα συμβαίνουν σε μια χώρα επηρεάζουν και τις άλλες ε, χώρες. Γι' αυτό ακριβώς όλοι μας πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο που θα μας επιτρέπει να συντονίζουμε τις ε, δράσεις μας και να διασφαλίζουμε ακριβώ αυτή την οικοδόμηση εμπιστοσύνη ε, μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων για να έχουμε μια βαθύτερη οικονομική και νομισματική ένωση. Ευχαριστώ. Έχουμε ένα αίτημα για το eye, Έχουμε δύο λεπτά για τον κάθε ομιλητή. Κύριος Ντάτμουθ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Έχω δύο πολύ απλές ερωτήσεις. Η πρώτη είναι. Υπάρχει πολύ υψηλή ανεργία των νέων στην Ισπανία. Και σε σχέση με το ερώτημα που έκανε ο προηγούμενος συνάδελφος, θεωρείτε ότι η μείωση του ελλείμματος του περιπολισμού είναι προς ε, το συμφέρον των εκατομμυρίων άνεργων, ειδικά άνεργων νέων. Και εάν ναι, ε, πώς μπορείτε να το θεωρείτε αυτό. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι πολύ απλά η εξής. Υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι στην Καταλωνία πρώην μέλη της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης της ε, Καταλωνίας και θέλει να τους ε, φυλακίσει η κυβέρνηση μέχρι και 25 χρόνια. Έχετε μια φήμη εσείς ε, ότι είστε υπέρ των ευρωπαϊκών αξιών. Προσωπικά λοιπόν πώς αισθάνεστε που είστε μέλος μιας τέτοιας κυβέρνησης που έχει πολιτικούς κρατούμενους και θέλει να τους φυλακίσει μέχρι και 25 χρόνια για καθαρά πολιτικούς λόγους. Πώς αισθάνεστε έτσι εσείς οι ε, λάτρεις ε, των ευρωπαϊκών αξιών. Θα ήθελα να τα ακούσω. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ντάτμουθ. Πρώτα απ' όλα για την ανεργία των ε, νέων. Έχετε απολύτως δίκιο. Είναι μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες και πρόβλημα, τα σημαντικότερα προβλήματα και πρέπει ακριβώς να προσπαθήσουμε να το λύσουμε το συντομότερο δυνατόν. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε ένα σχέδιο δράσης για τα ανεργία των νέων που θα χρησιμοποιήσει νομίζω πολύ καλά τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα εθνικά κονδύλια για να προσπαθήσει να δώσει ένα μέλλον σε όλους αυτούς τους νέους. Μειώνεται η ανεργία και είμαι σίγουρο ότι θα συνεχίσει και τους επόμενους μήνες, αλλά θέλουμε να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Αυτό βέβαια τελικά σημαίνει διαφορετικές δεξιότητες, εκπαίδευση κτλ. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε μέσω μακροπρόθεσμα, αλλά είμαι αισιόδοξη ότι ε, οι δουλειές οι οποίες ε, δημιουργούνται δεν είναι τόσο πολύ στον τομέα των κατασκευών, αλλά σε άλλους ε, κλάδους. Για το δεύτερο ζήτημα διαφωνώ δεν υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι στη χώρα μου. Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι είναι στη φυλακή γιατί παραβίασαν τους υφιστάμενους κανόνες. Αυτή είναι η πιο σαφής απάντηση στην πολύ έτσι, έντονη ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κανείς δεν αμφισβητεί το ότι η Ισπανία είναι κράτος δικαίου. Σας ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ. Ήταν εξαιρετικά θετικός ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων. Οφείλω να πω ότι ο προπολογισμό αυτός δείχνει το πώς είναι δυνατόν να συμβιβάσουμε την δημοσιονομική ευθύνη και μια όθηση στην κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη και πολλοί θα έπρεπε να δεχτούν από αυτό και η χώρα μου και η άποψή σας επίσης για την εμβάθυνση της ε, ΟΝΕ και την προτίμηση για την ε, κοινοτική μέθοδο και την ανάγκη για αυτήν τη λειτουργία σταθεροποίησης ε, νομίζω είναι πράγματα τα οποία καλωσορίζουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναμένουμε την συνεργασία μαζί σας με το Συμβούλιο και ελπίζουμε η διαδικασία η οποία ξεκίνησε να αποδώσει κάποια συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα για το νόμισμά μας αλλά και για τους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Yes. Yeah, colleagues, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν περάσουμε στις ε, ψηφοφορίες, ε, έχω δυστυχώς κάποιες ανακοινώσεις. Ε, αυτό είναι τα άσχημα νέα. Τα θετικά νέα είναι ότι η ψηφοφορία δεν θα κρατήσει πολύ. Είμαστε σύντομοι, αποτελεσματικοί. Είναι λίγες οι ψηφοφορίες. Οπότε μην ανησυχείτε. Θα κάνω λοιπόν κάποιες ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα λοιπόν οι γνωστές ανακοινώσεις του Προέδρου. Προπαρασκευαστική συνεδρίαση για τον επόμενο νομισματικό διάλογο που θα λάβει η χώρα στις 28 Ιανουαρίου 2019 θα είναι ο τελευταίος νομισματικός διάλογος αυτής της θητείας σας υπενθυμίζω ότι για να τιμήσουμε την 20η επέτειο του ευρώ θα έχουμε ένα μόνο θέμα όπως συμφωνήσαν οι συντονιστές, μια κριτική αξιολόγηση του εγχειρήματος του ευρώ όσον αφορά την αξιοπιστία, τη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και την στήριξη στο πλαίσιο της Νομισματικής Ένωσης. Προσκαλείστε όλοι με έξι ειδικού στην συζήτηση από το University College Dublin, τον Νοσά, το ΣΕΠΣ, το Ινστιτούτο του Κιέλου, το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και το ΕΛΕΣΥ. E. Θα συζητήσουν αυτά τα ζητήματα με τους ευρωβουλευτές. Θα λάβει χώρα Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019, μία με δυόμιση και θα μεταδοθεί στο διαδίκτυο. Τώρα, Έχουμε την ε, σύνοψη των συστάσεων ε, και των αποφάσεων των συντονιστών όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καμία γνωμοδότηση. Συμφωνήσαμε να καλέσουμε τους εκπροσώπους των εποπτικών αρχών ε, για να συζητήσουμε τα ζητήματα λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων για το θέμα του Δημοσιονομικού Συμφώνου θα, δεν θα ζητήσουμε γνωμοδότηση της Γιούρη για την εξέταση των επενδυτικών εταιριών. Έχουμε την ε, επιστολή της ΕΣΜΑ για το σκανδαλο κουμ CUM-X. Οι συντονιστές ήταν υπέρ του να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή να ερευνήσει το ζήτημα. Να... Συμφωνήσαμε όμως να μείνουμε το αποτέλεσμα του ψηφίσματος ε, της Ολομέλειας. Μετά έχουμε τα ζητήματα οικονομικής διακυβέρνησης, ε, την ε, Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα, την πρώτη συζήτηση είχαμε τα θέματα φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας, στην δεύτερη συζήτηση είχαμε την Τραπεζική Ένωση, το πακέτο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και είπαμε ότι ο οικονομικός διάλογος θα καλύψει και την περίπτωση της ε, Ιταλίας. Ε, επίσης συμφωνήσαμε να προσκαλέσουμε τον Υπουργό 3 και επίσης να υπάρξει μια συνεδρίαση για να εξετάσουμε τα πρίψε τον Φεβρουάριο 2019 αλλά μετά αποφάσισε να υπάρξει η ε, έκτακτη διαδικασία να υπάρξει δηλαδή μια δήλωση για την οδηγία για τη φεργιότητα υπαριθμών 2 την οποία θα σας διαβάσω σε λίγο αλλά πριν από αυτό καλωσορίζω και την Κομισιόν. Ναι, ναι, ναι, και η ΟΠΑ και τα λοιπά. Έχουμε λοιπόν την αναφορά από τις συνεχιζόμενες διοργανικές διαπραγματεύσεις τριμερής διάλογος για τις αποκαλύψεις στο θέμα των βιώσιμων επενδύσεων. Πρώτος γύρος έλαβε χώρα στο Στρασβούργο, στο είχαμε ακριβώ να δούμε τις διαφορές μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να καθορίσουμε το πεδίο της εφαρμογής όσον αφορά εταιρείε και προϊόντα, να επικαιροποιηθούν οι ορισμοί του κινδύνου, της αηφόρου επένδυσης, της δέουσας επιμέλειας, του συμμετέχοντος στην αγορά, του πιστοτικού ιδρύματος και είναι μια πρώτη συζήτηση για τις πράξεις κατεξιοδότηση. Συμφωνήσαμε ο επόμενο τριμερή διάλογο να γίνει στι 28 Ιανουαρίου. Για τα καλυμμένα ομόλογα είχαμε συνάντηση τριμερού διαλόγου στι 15 Ιανουαρίου. Μιλήσαμε ακριβώ ε, για τα καλυμμένα στοιχεία ενεργητικού και την ομοιογένειά τους. Ζητήσαμε από την Κομισιόν να συντάξει non-papers για αυτά τα ζητήματα και συμβαστικά κείμενα και για άλλα πολιτικά θέματα όπως παραδείγματο χάρη τις ε, κοινέ ε, ενδοομιλικές ε, δομές, την γενή χρηματοδότηση, τις απαιτήσει κάλυψης και ρευστότητας. Μετά έχουμε τον πρώτο ημερή διάλογο για τη συγκριτική αξιολόγηση 16 Ιανουαρίου για τους ορισμούς ε, για, τις, ε, για τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης ε, για την κλιματική μετάβαση, για τους στόχους των Παρισίων, για τις συγκεκριμένες απαιτήσει για την βιώσιμη ανάπτυξη. Ο επόμενος γύρος λοιπόν προβλέπεται για τις 30 Ιανουαρίου. Είχαμε και τον πρώτο τριμερή διάλογο για τον ΕΜΙΡ 2 και εκεί πέρα είχαμε εντατικές συζητήσεις ε, με τους συνομοθέτες ε, όσον αφορά το νέο καθεστώς για την εποπτεία ε, επενδυτικών σχημάτων τρίτων χωρών και την κατάταξή τους στην κατηγορία Tier 2 και την άρνηση αναγνώρισης. Δόθηκε εντολή στην Κομισιόν να συντάξει ένα non-paper το οποίο θα περιλαμβάνει πιθανώς και συμβαστικά κείμενα για την διάσταση των τρίτων χωρών, ενώ η διάσταση της ρύθμισης που αφορά τα ευρωπαϊκά επενδυτικά σχήματα δεν ε, μας απασχόλησε λόγω έλλειψης χρόνου και δόθηκε μια εντολή για προκαταρκτικές τεχνικές εργασίες. Και τώρα, όπως σας υποσχέθηκα, για την πράξη κατεξιοδότησης ε, για την φερεγγιότητα αποφάσισαν να κάνουν μια δήλωση οι συντονιστές προς την ΕΙΟΠΑ και προς την Κομισιόν. Καλωσορίζω την Ναταλή Βεζιέ, την επικεφαλής της μονάδας ε, από την ΕΙΟΠΑ και την κυρία Μίλλερ. Οπότε, εξ ονόματος της Επιτροπής μας θα διαβάσω τις ε, ανακοινώσεις αυτές για τον κανονισμό που τροποποιεί τον ε, δεύτερο κανονισμό για τις απαιτήσει κεφαλαιακής επάρκειας θα έπρεπε να έχει εγκριθεί το Δεκέμβριο του 2018, αλλά προετοιμάζεται ακόμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε. Άρα, αλλά ελπίζουμε ότι αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν αναλύει δεόντως και λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες μας και αναμένουμε να τα δούμε αυτά στην πράξη κατεξιοδότηση. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω τις ανησυχίες αυτές. Πρώτα απ' όλα, όπως αναφέρουμε στις επιστολές μας, θα θέλαμε να επαναλάβουμε την στήριξή μας για την μείωση του υφιστάμενου περιθωρίου κινδύνου για να χρηματοδοτηθεί η πραγματική η οικονομία και να υπάρξουν επενδύσεις σε μακροχρόνια έργα. Δεύτερον, αν και αναγνωρίζουμε ότι κάποιε από τι προτάσει μα για μια νέα κατηγορία επενδυτικών εργαλείων για μακροπρόθεσμε επενδύσει, έχουν υιοθετηθεί στο σχέδιο πράξη κατεξοδότηση, ανησυχούμε ότι όπω έχουν σχεδιαστεί αυτή τη στιγμή τα κριτήρια, όπω παραδείγματο χάρη είναι η 12 διάρκεια και η απαιτήσει περί ε, σημαίνει ότι ίσως δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει στην πράξη η νέα αυτή κατηγορία. Μάλιστα, όσον αφορά ακριβώς ε, το περιθώριο και τα νέα κριτήρια, αυτά θα μπορούσαν να επηρεάζουν σημαντικά τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και οι τροποιημένοι κανόνες ε, θα συνεισφέρουν στο να επιτύχουμε τους στόχους της Ένωσης των Χρηματαγορών με το να αφαιρέσουν τα υφιστάμενα εμπόδια στις ε, επενδύσεις ε, και τις επιχειρήσεις. Ε, τρίτων. τονίζουμε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ζητήσαμε από την Κομισιό να αναζητήσει λύσεις με βάση το εξτάμενο άρθρο 77 Δέλτα 4 της Οδηγίας Περιφερεγγιότητας, σύμφωνα με το οποίο συμφωνούν ο, οι νομοθέτες ότι θα πρέπει το εθνικό στοιχείο να ενεργοποιείται όταν πληρούνται τα κριτήρια στο τέλος της περίοδου και ανα πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της περίοδου αναφοράς με βάση καθημερινό υπολογισμό. Θεωρούμε λοιπόν ότι η πρόταση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με την οδηγία και σύμφωνη με τις αρμοδιότητες της ε, Κομισιόν για την πράξη κατά εξοδότηση. Τέλος, υπό το φως της καθυστέρησης ε, στην έγκριση της πράξης κατεξιοδότηση ανησυχούμε για το ότι η τωρινή ημερομηνία εφαρμογής μπορεί να, σημειώ... να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές δυσκολίες ε, δεδομένου του πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος θα περάσει μεταξύ της θέσεως ενισχύ και της πρώτης εφαρμογής για τις υποχρεώσεις αναφοράς. Η θα πρέπει να μειώσει τις αρνητικές συνέπειες για τις εταιρείε που θα συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη ε, το ότι έχουμε ήδη καθορίσει στόχους και προϋπολογισμούς. Ζητάμε από την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τις ε, συνέπειες ε, που θα προκύψουν όσον αφορά τις αναφορές ε, με βάση τι νέε διατάξεις και ειδικά με βάση τα υποδείγματα που θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό. Για όλα τα ανωτέρω θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό να περιμένουμε και προτείνουμε να εξεταστούν ε, στην έκθεση του 2018 μάλιστα εφόσον αναμένουμε τις αλλαγές ε, στο σχέδιο της πράξης κατεξοδότηση λυπούμαστε για το ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι οι περισσότερες προτάσεις της Επιτροπής μας ε, θα ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση της ε, εξέτασης οδηγίας για το 2020. Οπότε για να είναι ομαλή η διαδικασία ελπίζουμε η Κομισιόν να θελήσει να αξιολογήσει το πώς θα αντιμετωπιστούν οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου σε αυτή την πράξη του την πράξη κατεξιοδότηση και υπενθυμίζουμε εδώ πέρα το ότι έχει κάποια προνόμια σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης ε, το Κοινοβούλιο. Προνόμια τα οποία σκοπεύουμε να ε, ασκήσουμε και να εκμεταλλευτούμε πλήρως το σημαντικό αυτό νομοθέτημα. Και αυτό σημαίνει και την απόρριψη. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την υπομονή σας ήταν σημαντική νομίζω αυτή η δήλωση. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στις ε, τελευταίες ε, ψηφοφορίες. Ναι, ωραία, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, να κάνουμε ένα τεστ, μια δόκιμη. άρχια τη ψηφοφορία. Δουλεύει κύριε Γκέρερο, ωραία. Yes. So, uh, e, one EPP too many, sorry. Ε, είναι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Για ξαναπατήστε, παρακαλώ. Είδα έναν παραπάνω από το ΕΛΚ. Πρέπει να επαναλάβουμε το τεστ για να είμαστε σίγουροι. Πέρας. Τώρα. Θα δούμε. Ωραία, σας ευχαριστώ. Ξεκινάμε με την ψήφιση της προσωρινής συμφωνίας για την ελάχιστη κάλυψη απαιτήσεων για μη εξυπηρετούμενες ε, απαιτήσει ε, με ονομαστική ψηφοφορία, αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. 42 υπέρ, 10 κατά. Καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον συνεισηγητή και τώρα περνάμε στην έκθεση του κυρίου Σέλο για τον ΦΠΑ τροπολογίες 35 και 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 με προφορική τροπολογία από το ECR υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται οπότε ψηφίζουμε χωρίς προφορική τροπολογία υπέρ κατά νομίζω ίδια πλειοψηφία αλλά ας το δούμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 25 προς 26 Απορρίπτεται όμως. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας απορρίπτεται 48 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε και τη 48 πέρας απορρίπτεται 49 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε άρχιτη ψηφοφορία ψηφοφορία Μάλιστα. Ωραία, όλοι υπέρ ήταν. Λάθος, λάθος, δικό μου. Εγκρίνεται ομόφωνα λοιπόν. Αυτό, αυτό ήθελα, ναι. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 σε δύο μέρη, μέρος πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ, κατά να το επαληθεύσουμε. Πέρας. Η 52 καταπίπτει λοιπόν. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε την 62 άρχεται η ψηφοφορία και πέρασε απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά 70 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία 69 και 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 71 και 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε άρχιε την ψηφοφορία και πέρασε απορρίπτεται 20 με προφορική τροπολογία της ALDE υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ καταπίπτει συγγνώμη 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4, 4 είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 25 άρχεται η ψηφοφορία και πέρας. Εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 και 28 υπέρ, κατά, να την επαληθεύσουμε. Πέρας, εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 30 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 30. Πέρας. Απορρίφεται. Τι ήταν αυτό? 31 με προφορική τροπολογία. Υπέρ Κατά. Να την επαληθεύσουμε. Την 31. Προφορική τροπολογία. Πέρας. Απορρίπτεται. 31 χωρίς προφορική τροπολογία υπέρ. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, για την πρόταση της Κομισιόν όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Και πέρασε. 42 υπέρ, κανένας κατά, 10 αποχές, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνάμε τώρα. Στο επόμενο θέμα που είναι γνωμοδότηση του κύριου Φρουντζουλίκα. Απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών Συμβαστική Α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αναελέγξουμε. Ωραία. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίθηκε. 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, να ελέγξουμε. Τέλος, απορρίφθηκε με μικρή, πολύ μικρή διαφορά, καλά κάναμε και ελέξαμε. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε με μία ψηφοδιαφορά. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. 46 υπέρ, 2 κατά, 4 αποχές. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ίδιος εισηγητής τώρα, η ΕΙΟΠΑ. Συμβαστική Α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Γ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Δ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Ε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. 30 υπέρ 22 κατά εγκρίθηκε. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά κατά εσωλιστές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 19 ψηφίζουμε δε, ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίθηκε. 20. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25. Υπέρ κατά αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 25. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της υποφορίας. Απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. Ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. 44 υπέρ, 2 κατά, 4 αποχές. Εγκρίθηκε. Και περνάμε τώρα στην ΕΣΜΑ. Συμβαστική Α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Γ υπερκατά αποχές εγκρίνεται, Σεβαστική δέλτα, υπερκατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 9, υπερ, κατά, αποχές εγκρίνεται, αλλά θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος, εγκρίθηκε. 12 υπέρ, κατά,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 Ψηφίζουμε ολόκληρο το κείμενο, τροποποιημένο. Ψηφίστε παρακαλώ. Ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. 43 υπέρ, 2 κατά, 4 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Επόμενη συνεδρίαση Δευτέρα 28 Ιανουαρίου στις 3 και Τρίτη 29 το πρωί, 9 με 12.30. Σας ευχαριστώ πολύ. Έληξε η συνεδρίαση.